Ευχαριστώ. Τον, η συζήτηση έκλεισε και η ψηφοφορία θα γίνει στην πρώτη ολομέλεια του Μαρτίου. Προχωράμε τώρα στο επόμενο θέμα της εμερήσιας διάταξης που είναι η έκθεση από την κυρία Βάλαν σχετικά με τα ε, επενδυτικά προγράμματα για ενεργειακές υποδρομές στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και δίνω το λόγο πρώτα στην εισηγήτρια κυρία Βάλαν για δύο λεπτά. Για τέσσερα λεπτά, με συγχωρείτε. Thank you, Chair. And I fully appreciate... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκτιμώ ιδιαίτερα στην παρουσία σας. Επίτροπε και αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ όλους τους σκιώδεις εισηγητές για την συνεργασία τους η θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας δίνει στην Ένωση περισσότερες αρμοδιότητες στον ενεργειακό τομέα. Αυτό είναι ένας τομέας όπου εάν συνεργαστούν τα κράτη-μέλη θα έχουμε πιο ασφαλή και πιο φτηνή ενέργεια για τους πολίτες μας. Μαζί μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις ανεπιθύμητων γεγονότων όπως αυτά που συνέβησαν τον περασμένο χειμώνα. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε στη ροή φυσικού αραιίου εκτός των συνόρων μας ή να επιλύσουμε τέτοιου είδους διαφορές, αλλά μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η υποδομή μας θα καλύψει ελλείψεις και θα είναι πιο διαφανής και ξεκάθαρη η αγορά. Είναι μεγάλη προτεραιότητα το θέμα αυτό για την Ένωση. Έχουμε το τρίτο ενεργειακό πακέτο που υιοθετήσαμε πέρυσι για ένα πιο αποτελεσματική αγορά ενεργείας. Αυτή τη στιγμή εξετάζεται και άλλη μια πρόταση στο Ευρωκοινοβούλιο και αύριο θα συζητήσουμε και την ε, κανονισμό για την κοινοποίηση των επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα έτσι ώστε να γίνει πιο διαφανής η αγορά. Θα ήταν κρίμα λοιπόν με την ευκαιρία αυτή να μην χρησιμοποιήσουμε αυτό το νέο εργαλείο και να μην χρησιμοποιήσουμε την νέα νομική βάση που μας δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας το άρθρο 194. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό γιατί ο κανονισμός αυτός δεν είναι μόνο για να συλλέγει πληροφορίες αλλά μπορεί να δώσει μια γενικότερη εικόνα για τις υποδομές, για τις επενδύσεις στις ενεργειακές επίδομες. Αν λοιπόν το Συμβούλιο υιοθετήσει με λάθος νομική βάση τον κανονισμό αυτό, εγώ θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να προχωρήσει και να προσφύγει στο ΔΕΚ και σας διαβεβαιώ ότι θα το κάνει αυτό. Επί της ουσίας τώρα. Έχω ήδη πει στον κύριο Μπαρόζο και το λέω ξανά και εδώ σε εσά κύριε Επίτροπε ότι είναι σε καμπή η Ευρώπη και η προτεραιότητά μας τώρα θα πρέπει να είναι να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις μας και να δημιουργήσουμε ένα θετικό περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Χρειαζόμαστε ισχυρές πολιτικές και μια αξιόπιστη ενεργειακή πολιτική. Ο τελικός στόχος είναι να εξασφαλίσουμε φτηνή και ασφαλή ενέργεια και για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Με αυτή τη λογική ελπίζω ότι η συλλογή δεδομένων δεν θα γίνει αυτός σκοπός. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτός ο κανονισμός δεν θα δημιουργήσει άλλο ένα γραφειοκρατικό βάρος για τις επιχειρήσεις και ότι ο απόρριτος χαρακτήρας των ευαίσθητων πληροφοριών θα εφαρμοστεί. Για ένα άλλο θέμα. Λυπάμαι μόνο που το ΕΛΚ και η, ομάδα σοσιαλιστών και δημοκρατών εισηγάγαν μια τροπολογία που απαιτεί ευρωπαϊκές εταιρείες να δώνουν πληροφορίες για επενδύσεις σε τρίτες χώρες. Καλό οποιονδήποτε να μου πει ποια είναι η νομική βάση που να δίνει αυτή την εξοδαφικότητα. Επιπλέον, καλό θα είναι να ξέρουμε τι γίνεται πρώτα εντός της Ένωσης πριν κοιτάξουμε εκτός αυτής. Ξέρω ότι όλοι εδώ θέλουν να βάλουν τα πάντα σε αυτόν τον κανονισμό. Αυτό είναι λάθος πιστεύω. Για να είναι αποτελεσματικό αυτό το μέσο πρέπει να έχουμε συνεπείς πληροφορίες και να μην έχουμε υπερβολική γραφειοκρατία ούτε θέματα απορρίτου και για τις επιχειρήσεις μας και για την Κομισιόν. Προσπάθησα να βρω μια ισορροπία και δίνουμε την ευκαιρία στην Κομισιόν να κάνει μια αναθεώρηση μετά από πεθανές μελλοντικέ εξελίξεις αλλά να εξασφαλίσουμε ότι η εικόνα που θα έχουμε θα είναι ακριβής. Επίσης χρειαζόμαστε βεβαιότητα για μελλοντικέ επενδύσεις για να έχουμε καλή πολιτική και πρέπει να με καθησυχάσετε Επίτροπε ότι Θέλω να αποφύγω η Κομισιόν μετά την συλλογή των δεδομένων να αρχίζει να επιβάλλει επενδυτικά προγράμματα και να καταλήξει να λέει στις επιχειρήσεις το πού πρέπει να επενδύσουν. Πάντως πρέπει να δώσει λύσεις και κίνητρα έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να κάνουν βραχυπρόθεσμοι και μη κερδοφόρες επενδύσεις που ίσως χρειάζονται για την ασφάλεια των προμηθειών. Σταματώ εδώ. Σας ευχαριστώ και αναμένω τα όσα θα μας πείτε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Επίτροπος. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία ε, ε, Ισηγήτρια, κυρίες και κύριοι, η ενεργειακή κρίση πέρυσι έδειξε πόσο σημαντικό είναι να έχει η Ευρώπη μία ενεργειακή υποδομή η οποία δεν θα εξασφαλίζει μόνο την ε, λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αλλά θα μπορεί να βοηθήσει τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες σε περίπτωση κρίσεως. Γι' αυτό πρέπει να έχει μία επισκόπηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για το τι επενδύσεις προβλέπονται ή ε, ποιες εγκαταστάσεις παροπλίζονται. Γι' αυτό και προτείναμε να υπάρξει ένα νέο εργαλείο το οποίο θα πρέπει ε, να επιτρέψει να, τη λειτουργία σε περίοδο κρίσεως με τον τρόπο όπως λειτουργήσε το σύστημα στην πρώτη πετρελαϊκή κρίση. Και εδώ αναφέρομαι περισσότερο στις ανανεώσιμες πηγές ε, ενέργειας. Ε, χαιρετίζουμε τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για θέματα όπως την ε, ε, συμμετοχή ε, του αερίου, του άνθρακα, της θερμότητας και όλα τα θέματα Ωραία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους τεχνικούς. Οπότε κύριε Επίτροπε, αν θέλετε, μπορείτε να συνεχίσετε από το σημείο που είχατε διακόψει. Με ένα μικρόφωνο παρακαλώ. Μικρόφωνο παρακαλώ. Τώρα ναι. Λοιπόν, κύριε, κύριοι ε, ε, ε, Ευρωβουλευτές, είχα πει ότι όσοι βρίσκονται στην αίθουσα οι οποίοι ε, λαμβάνουν μετάφραση μπορούν να μου πούν ότι το σύστημα λειτουργεί να σηκώσουν το χέρι τους δηλαδή αντιλαμβάνουμε ότι τώρα το σύστημα λειτουργεί με συγχωρείτε κύριε Επίτροπε μήπως μπορείτε να ξαναξεκινήσετε και να δούμε αν μπορεί να υπάρξει μετάφραση και από τα γερμανικά κύριε Επίτροπε κύριε ε, Ευρωβουλευτέ είχα θέσει το ερώτημα πώς Υπάρχει κάποιο πρόβλημα καταφανώς με τα πολωνικά στο κανάλι 2 αντί για τα αγγλικά. Ε, Από αγγλικά αντιλαμβάνουμε ότι το σύστημα λειτουργεί. Τα γερμανικά λειτουργούν. Για να δούμε τώρα λειτουργεί το σύστημα. κύριε Επίτροπε, με συγχωρείτε και πάλι. Θέλετε να κάνετε άλλη μία προσπάθεια και ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά το σύστημα θα λειτουργήσει κανονικά. Κυρία Πρόεδρε. Είχα θέσει το ερώτημα ε, πώς ε, ε, θα αξιολογήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα δεδομένα που θα μας δώσουν τα κράτη-μέλη διότι ουσιαστικά θα πρέπει να προσαρμοστούμε ή στις ανάγκες της ζητήσεως και να δούμε αν μπορούμε να ανταποκριθούμε στα προγνωστικά ή προβλέπουμε θα υπάρξουν κενά. Είναι όμως ε, προφανές ότι σε σχέση με το ισχύον σύστημα ένας διάλογος στον τομέα αυτό θα πρέπει να βοηθήσει η θεσμικά και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει καταρχήν κάθε δύο χρόνια να καταρτίζει μία έκθεση σχετικά με τις διαρθρωτικές ε, εξελίξεις στις ενεργειακές υποδομές κατά τρόπον ώστε να υπάρξει βελτιωμένη ε, διαφάνεια σε όλους τους τομείς αυτής της αγοράς και να ξεκινήσουμε μία συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, τα κράτη-μέλη και να καταλήξουμε σε συμπεράσματα και τονίζω ιδίως αυτό το τελευταίο σημείο διότι είναι προφανές ότι ε, το, ο κανονισμός ε, προσπαθεί απλώς να συγκεντρώσει τα στοιχεία και να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες πώς θα διεκπαιρεώσουμε περαιτέρω τα θέματα στα πλαίσια μιας ε, συνεκτικής ενεργειακής περιοχής ακόμη είναι κάτι που πρέπει να καθοριστεί. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας θυμίσω το καινούριο άρθρο 194 της Συνθήκης Λισαβόνας που θα χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση αυτή. Το άρθρο αυτό για όλους μας, για το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μία ευκαιρία αλλά και μία υποχρέωση η ενεργειακή πολιτική να μπορέσει να διαμορφωθεί από κοινού με συμμετοχή όλων. Εδώ λοιπόν σε όλα τα νέα πολιτικά μέτρα θα πρέπει εγκαίρως να υπάρξει εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων και το νομοθέτημα στο οποίο βασίζεται η τωρινή συζήτηση αποβλέπει μόνο στη συγκέντρωση των πληροφοριών και κατά τη νομική άποψη της Επιτροπής βασίζεται σε τα άρθρα ε, ε, του, της συνθήκης Ευρατών και ε, θα πρέπει να επιλεγεί η νομική βάση, δηλαδή το δευτερογενές δίκαιο και συγκεντρώνοντας ε, τις πληροφορίες δεν μπορούμε να καταρτήσουμε μία ενεργειακή πολιτική γι' αυτό και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας από αυτού του σημείου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για την υπομονή σας με τα τεχνικά μας προβλήματα και τώρα απευθύνομαι στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και καταρχήν τον κύριο Μαρινέσκο ονόματι του ΕΛΚ για δύο λεφτά. Κύριε Επίτροπε, προσπαθήσατε να εξηγήσετε τον λόγο για τον οποίο δεν βρισκόμαστε σε συναπόφαση. Εγώ όμως συμφωνώ με την κυρία Βαλόν, την εισηγήτρια. Συμφωνώ μαζί της ότι θα ήταν καλύτερα να συζητήσουμε τον κανονισμό αυτό με διαδικασία συναπόφασης. Είναι πολύ σημαντικό νομοθετικό εργαλείο για την ενεργειακή αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θα πρέπει να συμπληρώνει μια εθνική και περιφερειακή ανάλυση και θα πρέπει να παγιώνει τις ενεργειακές πολιτικές μας να βρούμε τα κενά, τους κινδύνους σε ό,τι αφορά τις διάφορες δομές, τις επενδύσεις για να έχουμε ισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς. Νομίζω ότι η προσέγγιση της Κομισιόν έχει κάποια ασαφή σημεία τα οποία επιλύσαμε μέσω των τροπολογιών μας. Παραδείγματος χάρη η δημοσιοποίηση των στοιχείων που στέλνουν τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δημοσιεύονται και να είναι συνεπεί σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για να αποφευχθεί εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών. Και τι λέμε όταν λέμε ιδιαίτερος φορέας θα πρέπει να είναι ένας φορέας που υιοθετεί πολιετή επενδυτικά προγράμματα σε κοινοτικό επίπεδο. Θα πρέπει να αποφύγουμε, να αποφύγουμε επικαλύψεις σε ό,τι αφορά τη συλλογή όλων αυτών των στατιστικών στοιχείων και δεδομένων. Και ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η παρακολούθηση σε τρίτες χώρες παρακολούθηση των, Ευρωπαίων, των ευρωπαϊκών επενδύσεων που επηρεάζουν την ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά. Νομίζω ότι οι επενδύσεις σε τρίτες χώρες, οι κρατικές επενδύσεις και οι επενδύσεις που κάνουν εθνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να αναφέρονται αυτές αυτές και θα πρέπει στον κανονισμό αυτό να έχουμε μία νομική βάση. Ο κύριος Γκίρεκ. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση απαιτεί ασφάλεια και κοινή δράση στις επενδύσεις των κρατών μελών για τις ενεργειακές υποδομές σε όλα τα δίκτυα και για την ασφάλεια των επενδύσεων και τη διάθεση πληροφόρησης για τις υπάρχουσες εθνικές υποδομές, ενεργειακές υποδομές. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο ανταγωνιστικότητας στην αγορά υπηρεσιών και παραγωγής. Υπάρχει επίσης και το θέμα της εμπορικής μυστικότητας που δεν θα πρέπει να διακυβευτεί. χρειάζεται και η διαφύλαξη στρατιωτικών μυστικών. Τώρα για τους αγωγούς τύπου South Stream χρειάζεται να μην υποσκαφθούν τα συμφέροντα των κρατών μελών. Χρειάζεται συνεργασία, εμπιστοσύνη, αλληλεγγύη. Ο κανονισμός που προτείνεται μόνο μερικός ανταποκρίνεται σε αυτό το αίτημα. Θα πρέπει να ενσωματωθεί από τις προτεραιότητες των κρατών μελών. Η κυρία Εκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερος που είδα την δέσμευση εδώ της Κομισιόν να προωθήσει τις βέλτιστες πρακτικές και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της ενεργειακής αγοράς στην Ευρώπη. Αυτό είναι απαραίτητο και για τις θέσεις απασχόληση και την ανάπτυξη της Ευρώπης και είναι απαραίτητο να σεβαστούμε το όριο των δύο βαθμών Κελσίου. Έχοντας αυτά κατά νου πρέπει να έχουμε πιο αποτελεσματικά ενεργειακά δίκτυα και πιο αποτελεσματική εσωτερική ενεργειακή αγορά και αυτό απαιτεί η Κομισιόν να γνωρίζει τι συμβαίνει σε αυτή την αγορά και αυτό είναι στην ουσία το θέμα μας. Χρειάζεται όμως και η γριοφυκρατία που θα αντιμετωπίσει αυτή την πληροφορία. Δεν χρειάζονται επικαλήσεις. θα πρέπει οι πληροφορίες που χορηγούνται να είναι οι σκόπιμες για να επιτύχουμε τον στόχο μας. Αν θέλουμε πιο αποτελεσματική αγορά, τότε θέλουμε σημαντικές πληροφορίες από τις επιχειρήσεις, οι οποία όμως να διαπροστατεύονται και να μην παραβιάζεται το απόρριτό τους. Θα πρέπει να απορρίψουμε τις ε, τροπολογίες της ομάδας των πράσινων. Θεωρούμε ότι είναι τόσο σημαντική η πρόταση που θα πρέπει να έχει ως τομική βάση το άρθρο 195, δηλαδή να έχουμε μία τακτική νομοθετική διαδικασία σύμφωνα με αυτή τη συνθήκη. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι σωστή επιλογή και είναι μια κακή αρχή στην συνεργασία που χρειαζόμαστε με την Κομισιόν. Ένα λεπτό, κύριο Ζαντό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ καλό να συζητούμε αυτό το μέσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά το βασικό πράγμα για μας είναι η συναπόφαση. Μπορεί να είναι λοιπόν πιο αποτελεσματικό άμα πάρουμε συνολικά τις αποκεντρημένες ενέργειες. Δεν λέω εγώ να μετρήσουμε τον κάθε ηλιακό πίνακα αλλά θα πρέπει να γίνει η καταμέτρηση της αποκεντρωμένης ενέργειας και με να ακούω τη φιλελεύθερη συνάδελφο όταν μιλάμε εμείς για διαφάνεια να απαντάμε γραφειοκρατία. Πρέπει λοιπόν η Κομισιόν να διαβουλευθεί όλους τους ενδιαφερόμενους συνδικάτα και ενώσεις των κρατών μελών. Οι φορολογούμενοι συμμετέχουν σημαντικά στην προσπάθεια αυτής της μεταβατικής ενεργειακής περίοδου. Πρέπει όμως να ξέρουν σε προς ποια κατεύθυνση οι φορολογούμενοι χρηματοδοτούν αυτή τη μετάβαση και ελπίζω ότι θα ψηφιστεί ευρύτατα αύριο αυτό το μέτρο. Ο κύριος Στοσενόφσκι, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η ε, πληροφόρηση για τα ενεργειακά προβλήματα είναι αμφισβητήσιμη διότι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταγωνίζεται τις ιδιωτικές εταιρείε. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ε, ποιες είναι οι υποχρεωτικές πληροφορίες που πρέπει να δίδονται και το ο, ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών που θα πρέπει να διατηρείται. Ε, δηλαδή θα ε, επαρκεί να γνωρίζουμε περίπου τι δίκτυα πρόκειται να στο μέλλον και αυτό θα είναι ε, ικανοποιητικό και από εκεί και πέρα ε, μπορεί να δούμε εάν θεωρηθεί ότι δεν υπάρχουν επαρκείς επενδύσεις ή υπερβολικές επενδύσεις σε κάποιον τομέα. Ε, θα πρέπει κατά αυτόν τον τρόπο να αποφύγουμε και ορισμένες συζητήσεις για τα κρυφά σχέδια εταιριών. Κύριε Επίτροπε, οι εξελίξεις των τελευταίων ετών έδειξαν ότι δεν είναι πραγματικότητα η ασφάλεια των προμηθειών. Δεν είναι συμβατά τα συστήματα των κρατών μελών, ούτε επαρκώς συνδεδεμένα μεταξύ του. Πάντως πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκαν χωρίς φυσικό αέριο και χωρίς θέρμινση και δεν υπήρξε αλληλεγγύη. Για να διορθώσει αυτή την κατάσταση η Κομισιόν πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες και είναι λογικό λοιπόν να χρειάζεται πληροφορίες από τα κράτη-μέλη αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Για τους λόγους αυτούς πιστεύουμε ότι η πρόταση για ένα κανονισμό του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την κοινοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων είναι και απαραίτητη και φυσική. Ανταποκρινόμαστε λοιπόν στις εξελίξεις της ενεργειακής προμήθειας στην Ευρώπη. Οι τροπολογίες που υποβλήθηκαν ενισχύουν την πρόταση και θεωρώ ότι πρέπει να υποστηριχθούν. Με μονομένοι ομιλητές τώρα δεν φαίνεται εδώ η κυρία Σαρτόρη. Πρόεδρε, Πολύ σωστά η κυρία Μπαλνεάν στην έκθεσή της υποστηρίζει σημεία που εγώ συμμερίζομαι. Η... Τα στοιχεία τα οποία διαβιβάζονται είναι σημαντικότατα στοιχεία για τους διάφορους χρήστες, γι' αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε την ασφάλειά τους θα πρέπει να γίνει και σε περιφερειακό επίπεδο η καταγραφή. Επίσης η κοινοποίηση θα πρέπει να έχει και μία πρακτική σκοφιμότητα. Θα πρέπει να λειτουργεί ως συμπλήρωμα για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Θα πρέπει η Κομισιόν να τα διαπραγματευτεί όλα αυτά με τα κράτη-μέλη και το ανέλαβε αυτό ο Επίτροπος να το κάνει. Θέλουμε να αποφύγουμε επικάλυψη ε, της ε, ε, δουλειάς μεταξύ των ενδιαφερομένων, δηλαδή χρηστών, κρατών, μελών, περιφερειών και κομισιών για τη χρήση των δικτύων και αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα στην υποδομή για το φυσικό αέριο. Πρέπει επίσης να εγγυθούμε ότι αν οι χρήστες αλλάξουν σχέδια, επενδυτικά σχέδια δεν θα πρέπει να υποστούν πρόστιμα κανενός τύπου. Άρθρο 1 παράγραφος 2 τώρα της πρότασης όπου μιλάμε για το χρονικό περιθώριο της, για την προθεσμία κοινοποίησης. Πολλά σχέδια πολλές φορές παραμένουν μόνο στη φάση του σχεδιασμού. Καλό λοιπόν θα ήταν η κοινοποίηση να γίνεται μόνο για σχέδια εκείνα για τα οποία έχει δοθεί άδεια ή έχει ληφθεί η τελική απόφαση επενδύσεων. Η κυρία κυρια τικαου για ένα λεπτό τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εργασία της, γιατί η συνθήκη της Λισαβόνας ενισχύει την ε, θέση ε, της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής στο διομέα αυτό διότι μετά τις ενεργειακές κρίσεις είναι βασική πολιτική αυτή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για τα προγράμματα και τις επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα όπως και για ε, την ε, ε, αποθήκευση του αερίου θα πρέπει να αυξηθούν οι δυνατότητες και να επιζητηθούν λύσεις σε περίπτωση κρίσης δεν θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει μία επιπρόσθετη επιβάρυνση διοικητική στις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να επιβραβεύσει κανείς τις επιχειρήσεις οι ευρωπαϊκές οι οποίες επενδύουν σε τρίτες χώρες και επηρεάζουν την κατάσταση στις χώρες αυτές. Γι' αυτό και ελπίζω θα προσυπογράψετε την τροπολογία 74. Κύριος Χέλμερ, πολλές από τις τροπολογίες δείχνουν τη μανία μας για τις ανανεώσιμες. Μιλάμε για μείωση των εκπομπών ακόμα και αν η θεωρία της ανθρωπογενούς πρόκλησης της θέρμανσης του κλίματος καταραίει. Αλλά θα έπρεπε τότε να ήμασταν υπέρ της πυρηνικής ενέργειας και όχι των ανανεώσιμων. Και τώρα έχουμε κίνητρα που είναι υπέρ των ανανεώσιμων και κατά της πυρηνικής ενέργειας. Η Ευρώπη χρειάζεται ανταγωνιστική δυνατότητα παραγωγής ενέργειας που εύκολα επιτυγχάνεται με την πυρηνική ενέργεια. Δεν μπορούμε να βασιστούμε στις, στα αιωλικά πάρκα. Πολλές χώρες στην Ένωση, ακόμα και οι δικοί μου, αντιμετωπίζουν την δυνατότητα έλλειψης ενέργειας στο τέλος της δεκαετίας εξαιτίας της οδηγίας για τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εκτός και αν τελικά κατασκευάσουμε νέους πυρηνικούς αντιδραστήρες και νέα εργοστάσια αλλιώς θα σβήσουν τα φώτα. Ο κύριος Σόνικ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, τα ενεργειακά δίκτυα είναι βασικά θέματα για το μέλλον της Ευρώπης και η σημασία της ενεργειακής ε, τροφοδότησης είναι ένα βασικό σημείο που μας απασχολεί. Μετά όμως από αυτές τις δηλώσεις πρέπει να υπάρξουν στοιχεία για να μπορέσει να προχωρήσει η χρηματοδότηση. Η Exxon Mobile, μία από τη, ε, από τις μεγαλύτερες εταιρείες θεωρεί ότι ε, θα υπάρχει μία ε, αύξηση κατά 1,2% το χρόνο της απαιτήσεως κατανάλωσης πετρελαίου δηλαδή θα θέλουμε 35% περισσότερα μέχρι το 2040 προς το παρόν χρησιμοποιούμε δισεκατομμύρια κυβικών αερίου που επίσης θα αυξηθούν κατά 44% και κατόπιν αυτών των προοπτικών η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενεργειακή υποδομή θεωρείται στρατηγικό θέμα και είναι δύσκολο να βρει κανείς επενδυτές για διάφορα θέματα ε, και περαιτέρω ένα άλλο θέμα που θα επιτρέψει τις επενδύσεις είναι να προτιμήσει κανείς διασυνοριακά προγράμματα τα οποία συμβάλλουν και εις την βελτίωση της τροφοδότησης και ε, κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει κανείς να βελτιώσει ε, και τις ε, συγγενείς διεργασίες. Τώρα ξεκινά η διαδικασία ΚΑΤΣΤΙΑΗ καταρχήν με τον κύριο Κέι. Κέλλη. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για τρεις διαφορετικούς λόγους τι θα γίνει όταν δεν θα έχουμε πλέον ορυκτά καύσιμα για τις κλιματικές αλλαγές και τους στόχους μου του 2020 όπου ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ο στόχος μας θα πρέπει να είναι μείωση κατά 30% και τρίτον να μειώσουμε την εξάρτησή μας από ορεκτά καύσιμα που προέρχονται από μη δημοκρατικά καθεστώτα και ασταθείς περιοχές. Δεν έχουμε χρόνο λοιπόν και ένας τομέας που απαιτεί προσοχή είναι η έρευνα και η καινοτομία και εγώ ανησυχώ για πιθανή επικάλυψη στον τομέα αυτό. Πρόσφατα έμαθα ότι υπάρχουν 45 διαφορετικές ομάδες που διερευνούν τα βακτήρια της αλμονέλας. Θα μπορούσατε να είχατε 50 ομάδες για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε για ηλιακή ενέργεια είτε αιωλική. Οπότε ρωτώ την Κομισιόν πώς σκοπεύει να τα συντονίσει όλα αυτά για να χρησιμοποιήσει τους κατάλληλους πόρους για να επιτύχουμε την απαραίτητη τεχνολογία. Ο κύριος Ένσιου. Πρόεδρε, συγχαίρω την εισηγήτριά της για την έκθεσή της. Θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποια σημεία για την συνεχιζόμενη ανάπτυξη των ενεργειακών υποδομών. Αυτό είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τις αλλαγές που έχουμε μπροστά μας. Πρέπει να επενδύσουμε σε νέα δίκτυα προσαρμοσμένα στα νέα είδη ενέργειας. Αυτό είναι απαραίτητο για να έχει ο πληθυσμός πρόσβαση σε νέες μορφές ενέργειας. Αυτή τη στιγμή η περιφερειακή συνεργασία de facto υφίσταται, αλλά θα πρέπει να ενισχυθεί με ξεκάθαρους κανόνες και να υπάρχει αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη-μέλη η οποία θα πρέπει να είναι πραγματικότητα. Περισσότερη επένδυση για συστήματα πληροφορικής για παρακολούθηση των αποθεμάτων σε περιόδους κρίσεων. Τέλος, να σας πω ότι οι επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα και στην πληροφορική είναι πολύ καλές εξελίξεις για την μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Ο κύριος Νικολάσιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συνθήκη της Λισαβόνας ενισχύει ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτή η δυνατότητα για να αποφύγουμε περαιτέρω προβλήματα στον ενεργειακό τομέα. Το να δίδονται πληροφορίες για τις επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές θα επιτρέψει να εντοπίσουμε τα κενά μεταξύ προσφοράς και ζητήσεως και να μπορέσουμε καλύτερα να διαμορφώσουμε την κοινή πολιτική στον τομέα της ενέργειας και της σχετικής αγοράς. Γι' αυτό και θεωρώ ότι θα πρέπει από κοινού να συγκεντρώσουμε τις αναγκαίες πληροφορίες για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε την ενεργειακή πολιτική ε, βάσει των ε, ε, συστημάτων που υπάρχουν σε κάθε κράτος. Ευχαριστώ για την ενεργειακή προμήθεια ε, υπάρχουν προτεραιότητες και στα κράτη-μέλη αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει μια ιδιαίτερη ευθύνη η οποία πρέπει να εξασφαλίσει την ενεργειακή ασφάλεια ε, με την ε, αρμόζουσα εποπτεία του, της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Αγοράς. Στους μηχανισμούς αυτούς θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η στήριξη των πολύ αποτελεσματικών επενδύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα πρέπει να αναθέσει μελέτες οι οποίες θα βασίζονται σε αξιόπιστες ε, ε, υποδομές κράτη-μέλη και θα πρέπει να λάβει υπόψη της ότι θα χρειαστεί μεγαλύτερη διαφοροποίηση της προμήθειας ενεργείας, της ε, μεταφορέας και των πρώτων υλών. Ε, μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να διατυπώσει την καλύτερη στρατηγική για την Ευρώπη η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Ρούμπικ. Πρόεδρε. Ένα από τα βασικά θέματα εις ε, την ενεργειακή πολιτική είναι ε, ε, ο τρόπος αποθήκευσης και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποθηκεύσουμε περισσότερο ενέργεια, πράγμα που είναι μεγάλη πρόκληση και για τις νέες ενέργειες. Χρειαζόμαστε όμως πιο έξυπνα δίκτυα, διότι όσο περισσότερη ενέργεια έχουμε, τόσο περισσότερο εάν έχουμε έξυπνα δίκτυα θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε τον κόσμο μας και τέλος θα πρέπει να θέσουμε κίνητρα στους προπολογισμούς να μειώσει κανείς το κόστος ε, στους ε, προϋπολογισμούς των διαφόρων χωρών. Για το μέλλον νομίζω ότι όλα αυτά θα έχουν μεγάλη σημασία στο μέλλον, όχι μόνο για την ε, παραγωγή αλλά και για την κατανάλωση ενέργειας. Σας ευχαριστώ. Και τώρα δίνω το λόγο στην Επιτροπή, στον Επίτροπο. Äh, Κυρία <coughs> Πρόεδρε, κύριε ε, Ευρωβουλευτέ, σας ευχαριστώ για τις χρήσιμες ε, υποδείξεις, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα, θα λάβει υπόψη της την τελική μορφή των προτάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά το σχετικό κανονισμό, διότι ε, γνωρίζετε ποια είναι τα προγράμματά μας και συμφωνούμε με την πρόθεση να διατυπώνουμε και να δημοσιεύουμε στοιχεία μόνο εφόσον ενδιαφέρουν το σύνολο χωρίς όμως ε, να υπάρχουν παραπομπές σε μονομένες ε, επιχειρήσεις. Αυτή, αυτό το βασικό στοιχείο όπου θα πρέπει ε, κάθε φορά να εξετάζεται μόνο ένα επίπεδο της της ενέργειας είναι πολύ σημαντικό και ε, πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει εντός πέντε, πέντε ετών να έχουν διατυπώσει τα μεθόδους αποθήκευσης της ενεργείας και ο κανονισμός θα επιτρέψει μία μεγάλη συζήτηση στα θέματα των υποδομών διότι χρειάζεται και ε, ε, υποδομή αλλά και κάποιο όργανο αλληλεγγύης που να μπορεί να επεμβαίνει στα δίκτυα ε, όπως άλλωστε θα πρέπει να υπάρχουν και εκθέσεις προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του ενεργειακού προγράμματος. Σας ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Βάλε, ανησυγήτριά μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι για τη σημαντική σας συνεισφορά στη συζήτηση. Δύο λόγια μόνο ως το δικό μου συμπέρασμα. Τονίζω για άλλη μία φορά ότι οι πολιτικές δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουν στην αγορά. Μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη είναι πολιτική, είναι ελεύθερη αγορά και οι πολιτικές πρέπει να διορθώσουν τις αδυναμίες της αγοράς και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον κανονισμό για να έχουμε σωστή εφαρμογή άλλων κανονισμών ή να ζητάμε εξαντλητικές πληροφορίες. Δεν ζητάμε στατιστικά στοιχεία. Πρέπει να είναι σχετικές οι πληροφορίες γιατί αλλιώς δεν θα έχει κανένα σκοπό η συλλογή τους. Δεν κάνουμε πολιτική με τον κανονισμό αυτό για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή το φυσικό αέριο. Και τέλος, προς την κυρία Εκ, θα ήθελα να πω ότι ελπίζω ότι τα συνολικά δεδομένα μετά από αυτόν τον κανονισμό θα μας βοηθήσουν να γίνουμε πιο έξυπνοι σε ενεργειακά θέματα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. This debate is now closed and the vote will take place at 11:30 tomorrow. Ευχαριστώ. Η συζήτηση θα συνεχιστεί, ε, η συζήτηση έληξε και ε, η ψηφοφορία θα είναι αύριο Πέμπτη. Η επόμενη έκθεση είναι ε, του κυρίου Μάνκα σχετικά με την τροποποίηση της κατάστασης προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον